προσώπου για την κατάσταση στη Σαουδική Αραβία και στο Ιράν. Κυρία Μογκερίνη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρωτού περάσω στις λεπτομέρειες της κατάστασης, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα όσον αφορά τα όσα έγιναν στη Βιέννη το Σάββατο, όπου καταφέραμε να δείξουμε ότι ακριβώς έξι μήνες μετά την συμφωνία που υπογράψαμε με το Ιράν για το πυρηνικό τους πρόγραμμα, το Ιράν τελικά πληρεί τις υποχρεώσεις του και τις δεσμεύσεις του, τις οποίες είχε αναλάβει και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επαλήθευσε την κατάσταση αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις υπόλοιπες δυνάμεις, τις οποίες συντονίζω εγώ, επιβεβαίωσε και αυτή ότι όντως η συμφωνία υλοποιείται και ότι εφαρμόζεται από... Και ας θυμηθούμε ότι πριν από έξι μήνες υπήρχαν πάρα πολλοί, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά γενικότερα στην περιφέρεια, στην περιοχή εκείνη που εξέφραζαν έναν πολύ έντονο σκεπτικισμό σχετικά με το αν θα καταφέρναμε ποτέ όχι μόνο να υπογράψουμε συμφωνία, αλλά και να υλοποιηθεί η συμφωνία αυτή και μάλιστα πολλοί θεωρούσαν ότι το Ιράν δεν θα εκπληρούσε σε καμία περίπτωση τη συμφωνία αυτή και ότι δεν θα προχωρούσε σε συγκεκριμένε πράξεις για την υλοποίηση της συμφωνίας. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι ε, προφανώς μιλάμε αυτή τη στιγμή για διαπραγματεύσει που έχουν να κάνουν με ένα πυρηνικό πρόγραμμα και ικανοποιούμεθα ως προς αυτό το ότι ουσιαστικά αποφύγαμε το μεγάλο αυτό κίνδυνο της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και τον κατ' κίνδυνο μιας γενικότερης διένεξης στην περιφέρεια. Αυτό λοιπόν με ικανοποιεί ιδιαίτερεως, αλλά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο με ικανοποιεί και έχει να κάνει αυτό με το ότι δείξαμε ότι η πολυμέρεια, η διπλωματία, οι πολυμερείς σχέσεις πραγματικά λειτουργούν στην πράξη. Όχι μόνο για τις περιφερειακές όμως συμφωνίες, αλλά ότι μπορούν να αλλοποιηθούν και ως συμφωνίες οι οποίες λειτουργούν στην πράξη. Αυτό λοιπόν το βρίσκω ιδιαίτερα θετικό και περνώντας τώρα στην συζήτηση που προβλέπεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν δύο ακόμα ελπιδοφόρα στοιχεία. Το ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε καλύτερες διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Ιράν και του υπόλοιπου κόσμου, ξεκινώντας από τις σχέσεις μεταξύ Ιράν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαμε και εμείς ως Ευρωπαίοι να, μπορούμε, να συνεργαζόμαστε καλύτερα με το Ιράν πλέον σε πάρα πολλούς τομείς και Τέλος, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό ελπιδοφόρο στοιχείο είναι ότι η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικές σχέσεις γενικότερα στην περιοχή. Και έρχομαι τώρα στο ζήτημα το οποίο θα εξετάσουμε σήμερα το βράδυ. Γιατί ξέρετε ότι ε, καταφέραμε μέσω διαπραγματεύσεων που κράτησαν 13 ολόκληρα χρόνια με πάρα πολλές δύσκολες στιγμές, με πάρα πολλές διακυμάνσεις, με πάρα πολύ σκεπτικισμό. Καταφέραμε παρόλα αυτά μετά από τόσα χρόνια να καταλήξουμε σε μια ιστορική συμφωνία, άλλο των προβλέψεων θα και κανείς. Θεωρώ λοιπόν ότι ανάλογα θα πρέπει να καταβάλουμε παρόμοιες προσπάθειες προκειμένου να έχουμε μια διαφορετική θετική πλέον συνεργασία στην όλη αυτή περιοχή. Δεν είμαι αφελής, ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολο κάτι τέτοιο, ξέρω ότι δεν θα συμβεί εν μία νυχτή, αλλά σίγουρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία θα έρθουν μπροστά μας. Το γεγονός ότι θα υπάρξουν ορισμένοι που δεν θα θέλουν τελικά να συνεργαστούν για τα ζητήματα αυτά, αλλά νομίζω ότι ε, ήδη αυτή τη στιγμή έχει σημειωθεί μια σημαντική πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν. Θα αποτελήσει αυτό για μας μια πολύ σημαντική δοκιμασία, μόνο και μόνο η εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Αλλά σκεφτείτε πως είχε κατάσταση πριν από ένα χρόνο. Ορισμένοι πίστευαν δεν θα καταλήγαμε ποτέ σε συμφωνία με το Ιράν, ότι η συμφωνία αυτή δεν θα εφαρμοζόταν ποτέ. Αυτοί λοιπόν διαψεύστηκαν. Αν καταφέρουμε λοιπόν ενωμένοι ως Ευρωπαίοι να συνεργαστούμε με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, είμαι πεπισμένη ότι θα συνεχίσουμε να εκπλήσουμε με κάποιο τρόπο όλους αυτούς τους σκεπτικιστές. Ο διάλογο λοιπόν πρέπει να ξεκινήσει για όλε αυτέ τι περιφερειακέ δυνάμει, αρχή γενομένη από τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε τελικά να βγούμε από τη δύσκολη αυτή κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια ξέρετε ότι υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση όσον αφορά την επικράτηση, μια γεμονική επικράτηση στην περιοχή. Είχαμε αρχικά την ΝΤΑΕΣ, η οποία προσπάθησε ω οργάνωση να αποσταθεροποιήσει περισσότερο την περιοχή και να την οδηγήσει σε χάο. Είχαμε επίση και Διενέξει όπω είδαμε μεταξύ Σαουδική Αραβία και Ιράν και θα μπορούσαν και αυτέ οι διενέξει να ενταχθούν σε μια γενικότερη λογική θρησκευτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ Σουνιτών και Σιητών. Καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνο που ελοχεύει αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο. Μπορεί πραγματικά να τροχοπεδίσει την προσπάθεια ειρήνευσης ακόμη και στη Συρία. Εμπλέκεται το ζήτημα αυτό επίση και με το ζήτημα τη Ιεμένη που θα συζητήσουμε αύριο. Θα μπορούσε η διένεξη αυτή να αποσταθεροποιήσει και το ίδιο το Ιράκ, το Λίβανο, τις δύο αυτές χώρες στην περιοχή οι οποίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε εκταριστικό εξτρεμισμό, αλλά θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει η διένεξη αυτή σε τεράστια αποσταθεροποίηση ακόμα και της Ασίας και της Αφρικής και της γενικότερης περιοχής του Σαχέλ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να αναζωροποιηθεί η ένταση στην όλη περιοχή και τελικά να τροχοπεδίσει και πολλές άλλες προσπάθειες που γίνονται στην περιοχή αυτή και να οδηγήσει τελικά και σε μια γενικότερη παγκόσμια αποσταθεροποίηση. Γι' αυτό ακριβώς εμείς θέλουμε μια αποκλιμάκωση της έντασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχοντας ένα απόλυτο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι μαζί ενωμένοι θα πρέπει να στείλουμε το ίδιο μήνυμα και με τους διεθνούς μα εταίρους. Και φέρουμε προφανώς στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες δυνάμεις. Για παράδειγμα η Ινδονησία, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδονησίας με τον οποίο συναντήθηκα πριν από μερικές ε, ημέρες μου είπε και αυτός ότι θα καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της ε, έντασης στην περιοχή αυτή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι προσπάθειες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί ουσιαστικά επηρεάζουν ή ε, δυνητικά μπορούν να επηρεάσουν τρεις ή και τέσσερις υπήρους. Και καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές κοινότητες ανά τον κόσμο που θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε περισσότερη ένταση. Εμείς μετά τη, τα γεγονότα της Δευτέρας Ιανουαρίου και μετά την εκτέλεση του ΣΥΤ Μάμι Νίμρα Αλ Νίμρα από τις οδικές σαδραβικές ε, αρχές αναλάβαμε αμέσως δράση και επίσης αντιδράσαμε και κατά των ε, εκτελέσεων άλλων κρατουμένων που είχαν ε, καταδικαστεί από τη Σαουδική Αραβία για τρομοκρατία. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε εμείς να υποστηρίξουμε την θανατική αυτή ποινή δεν αποτελεί λύση για την τρομοκρατία. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν ήταν κατά της θανατικής ποινής οποιοδήποτε και είναι το αδίκημα και νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε αγώνα για την παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής. Βέβαια αυτό ισχύει και για το Ιράν, όπου ο απολογισμός της κατάστασης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα βέβαια δεν είναι πάρα πολύ θετικός και το μήνυμα αυτό έχει περάσει βέβαια και προς τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν αλλά και προς τον Υπουργό Εξωτερικών της Αδικής Αραβίας με τους οποίους ήρθα σε επαφή τις τελευταίες μέρες. Μας ενισχύει ιδιαίτερα η περίπτωση του Νίμρα Αλ Νίμρα της εκτέλεσής του. Είναι ένα ζήτημα μη προάσπισης της ανθρώπινης ζωής, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντάξουμε το ζήτημα αυτό και στην γενικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αντιδράσαμε μετά, τα όσα έλαβαν χώρα στο Ιράν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πρεσβειών. Γιατί είδαμε ότι στο Ιράν σημειώθηκαν πάρα πολλές επιθέσεις κατά της πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας Είπαμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το Ιράν να τηρήσει τις ε, διεθνείς δεσμεύσεις του και προφανώς να προστατεύσει σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε διπλωματική αντιπροσωπεία. Συνομιλώντας και με τις δύο πλευρές τηλεφωνικά, το βασικό μου μήνυμα και επίσης στις επαφές που είχαμε και μετά τις τηλεφωνικές αυτές επαφές, όπως σας είπα συναντήθηκα με τους αρμόδιους υπουργούς κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού, το βασικό μήνυμα πάντως που πέρασε σε όλες τις περιπτώσεις ήταν ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις διμερείς εντάσεις χωρίς να αναζωπυρώνουμε και να αναμοχλεύουμε τα πάθη σε όλη την περιοχή. Και είπα παράλληλα ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ειρήνευση τόσο στη Συρία όσο και στην Ιεμένη και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι δύο αυτές χώρες να αποσταθεροποιηθούν από τη διένεξη μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, όπως δεν θα πρέπει να αποσταθεροποιηθεί περαιτέρω το Ιράκ ή ο Λίβανος. Και είπε επίσης ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε πάση θυσία τις ειρηνευτικές αυτές διαδικασίες, τις διαδικασίες αυτές σταθεροποίησης. Μιλήσαμε πριν από λίγο για το ζήτημα της Συρίας, συντοποιούμε, αν δεν κάνω λάθο όλοι, ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να συμβάλλουν, πραγματικά θέλουμε ειρήνη στην περιοχή και για ακριβώς τον ίδιο λόγο ήδη από τις πρώτες μέρες του έτους αυτού συζήτησα με όλους τους ηθήνοντες τους κινδύνους για την, για την περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης. Συζήτησα με το Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών, καθώς επίσης και με ηγέτες και υπουργούς αραβικών, αφρικανικών και ασιατικών κρατών και αναλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή δράση όχι μόνο με τους εταίρους μας, αλλά κυρίως μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως άλλωστε φάνηκε και από το χθεσινό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Είπαμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση έκβαση διαπραγμάτευση στη Μέση Ανατολή γενικότερα και αυτό είναι προς το συμφέρον όλων μας και προφανώς προς το συμφέρον της περιοχής αυτής. Ο πόλεμος μόνο τους τρομοκράτες ευνοεί και ουσιαστικά προωθεί την αποσταθεροποίηση πέρα από τα όρια της Μέσης Ανατολής και στην Ευρώπη όπως το έχουμε δει τελευταία. Αυτό είναι το ισχυρό μήνυμα το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε προς το Ιράν και προς τη Σαουδική Αραβία. Και είναι πάρα πολύ σημαντική η ευκαιρία που μας δίνεται για να σταματήσουμε την ένταση στην περιοχή αυτή προκειμένου να σταματήσει και η περαιτέρω αποσταθεροποίηση σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. καταλαβαίνω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα αποφεληθούν όλε οι πλευρέ. Γιατί αν δεν υπάρχει μια λύση που να αποφελεί όλε τι πλευρέ, η λύση αυτή τελικά θα είναι το χάο, το διευρυμένο χάο. Ξέρετε ότι χρειάστηκαν να περάσει πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούμε μια ειρηνική συμφωνία για την Συρία. Βλέπουμε επίση ότι ε, αυτή τη στιγμή η διεθνή κοινότητα φαίνεται ότι θέλει να συμβάλλει για μια ειρήνευση στη Συρία. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν θα πρέπει να χάσουμε την θετική αυτή δυναμική που έχει δημιουργηθεί και σε καμία περίπτωση όλες αυτές οι χώρες της περιοχής δεν θα πρέπει να εκτεθούν περισσότερο αυτή τη στιγμή σε περισσότερο ένταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να κάνει κάθε το δυνατό για να προωθήσει το διάλογο, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας Γι' αυτό διότι έχουμε αντλήσει και εμείς κάποια σημαντικά διδάγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το είπα και στην προηγούμενη παρέμβασή μου, στο προηγούμενο σημείο της σημερινής διάταξης, όταν συζητούσαμε την περίπτωση της Κολομβίας. Συντοποιούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο ότι η περιφερειακή μόνο συνεργασία οδηγεί σε ειρήνη και σε ευημερία. Το έχουμε δει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, ότι μόνη η λύση αυτή τελικά μπορεί να λειτουργήσει και ότι μόνο κατά αυτόν τον τρόπο τελικά μπορούμε να δώσουμε τέλος στον πόλεμο και να εγγυηθούμε την ειρήνη. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να λειτουργήσουμε μόνο μέσω της περιφερειακής συνεργασίας και ποτέ μέσω του ανταγωνισμού ή της αντιπαράθεσης. Και αυτό ισχύει σίγουρα πολύ περισσότερο για την περιοχή αυτή του κόσμου, τη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Πρέντα έχει τώρα πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, η Σαουδική Αραβία και ορισμένοι Σουνίτες σύμμαχοι φίλοι της έχουν διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την Τεχεράνη στην αρχή της χρονιάς. Υπήρξαν διαδηλώσεις μετά την εκτέλεση ενός επικεφαλής Σιήτη ηγέτης της 2 Ιανουαρίου. Εκτέλεση 47 ατόμων κεφατισμό του σε είναι η πιο μεγάλη εκτέλεση που έχει κάνει ποτέ η Σαουδική Αραβία από το 1980. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι απορρίπτουμε τη θανατική ποινή με κατηγορηματικό τρόπο. Το είπατε και εσείς κυρία Μογκερίνη. Πρέπει να τηρήσουμε αυτή τη δέσμευση όλοι. Να μην ε, ξεχνάμε ότι ο απολογισμός του Ιράν ως προς τη θενατική ποινή δεν είναι καθόλου λαμπρός. Πέρσι, ενώ είχαν σημειωθεί πρόοδοι για τα πυρηνικά, στο Ιράν έγιναν 1084 εκτελέσεις και γι' αυτό χαίρομαι που στη σημερινή συζήτηση προσθέθηκε και το Ιράν, γιατί στην αρχική πρόταση των ε, αριστερών, κομμουνιστών, σοσιαλιστών και φιλελεύθερων φίλων μας ήταν να γίνει συζήτηση μόνο για τη Σαουδική Αραβία και να κριτικάρουμε μόνο τη Σαουδική Αραβία και όχι τους υπόλοιπους. Νομίζω λοιπόν ότι τώρα είμαστε μπροστά σε μια νέα φάση αντιπαλότητας Σιητών και Σουνιτών. Δυσκολευόμαστε να δεχθούμε το χάσμα μεταξύ των δύο. Είναι λάθος αυτό. Και πρέπει πολύ σοβαρά να λάβουμε υπόψη αυτά που μας είπε η κυρία Μογκερίνη. Δηλαδή να καταλαγιάσουμε αυτή τη σύγκρουση η οποία θα μας πλήξει με δραματικό τρόπο τα επόμενα έτη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάουιτ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε την εφαρμογή του κοινού περιεκτικού και ολοκληρωμένου σχέδιου δράσης και ο εισηγητή πρέπει να έχει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να έχουμε μια νέα συνεργασία με το Ιράν. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε κοινά συμφέροντα και με το Ριάντ και με την Τεχεράνη και στα ενεργειακά θέματα και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τώρα υπάρχει θέμα με τη θανατική ποινή, με τα δημοκρατικά πρότυπα, με τη δικαιοσύνη, με τις θρησκευτικέ μειονότητες και με τους περιορισμούς έναντι των γυναικών. Και οι δύο χώρες δεν πρέπει να δίνουν εξωτερική χρηματοδότηση που αποστοθεροποιεί και δεν πρέπει να στηρίζουν εξτρεμιστικές ομάδες. Ζητώ από την κυρία Μογκερίνη να μας πει ε, ε, ποια, θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, είναι πολιτικώς αντιφρονούντες, δεν είναι τρομοκράτες. Ο άμαχος πληθυσμός είναι στο στόχαστρο στην Ιεμένη και όλα αυτά αποτελούν παραβάσεις του κώδικα διοντολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι πετύχαμε να σταματήσουμε έναν αγώνα δρόμου για τα πυρηνικά στην περιοχή και τώρα χρειάζεται ίδια δράση και για τα συμβατικά όπλα. Ξέρετε, για αιώνες ε, συνυπάρχουν ειρηνικά Σιήτες και Σουνίτες. Πρέπει να σεβαστούμε τις διαφορές μέσα στο Ισλάμ που υπάρχουν εδώ και αιώνες, αλλά να έχουμε τη σωστή πολιτική συνεργασία για το μέλλον. Και το Ιράν και η Σαουδική Αραβία έχουν ρόλο να διαδραματίσουν στην περιοχή. Και δεν πρέπει το, για να έχουμε το ένα να πρέπει να θυσιάσουμε το άλλο. Και οι δύο χώρες μπορεί να είναι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο οι άλλοι κόβουν διπλωματικούς δεσμούς, εμείς θα πρέπει να τους εντείνουμε και να τους συσφίγγουμε. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να είμαστε ε, ε, ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας και η δημοκρατία του Ιράν δεν ε, συμβάλλουν θετικά στην ανθρωπιστική κατάσταση και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Ε, απέχουμε πολύ από τους στόχους μας. Οι τζιχαντιστές έχουν, είναι πολύ καλύτερα δικτυωμένοι και επίσης συνεργάζονται με τη Σαουδική Αραβία και με την Αλκάιντα όπως υπόθηκε εδώ. Δηλαδή οι υπηρεσίες πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται στο Ριάντ. Όσον αφορά το Ιράν θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τους τζιχαντιστές από κοινού με τη Σαουδική Αραβία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, αυτό το οποίο ενώνει τη Σαουδική Αραβία και το Ιράν είναι περισσότερο από αυτό που τους ε, χωρίζει. Ατιμορρησία, θεσμοθετημένη ε, βασανιστήρια, θεσμοθετημένα βασανιστήρια, αποκεφαλισμοί κλπ. Ε, πέρα από αυτές τις ε, εξερμιστικές ομοιότητες ε, υπάρχει και μια άλλη σημαντική ομοιότητα, το πετρέλαιο και ε, το λαθρεμπόριο πετρελαίου παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το γεγονός ότι το Ιράν εγκαταλείπει το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι θετική ένδειξη για την ειρήνευση, αλλά δεν μπορεί να είναι άλοθη για να αμβλύνουμε τις απατήσεις μας όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την άσκηση επιρροής, ούτε ώστε η Ιρανική κυβέρνηση να εκπληρώνει τα, να πληρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όσον αφορά τις σχέσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράν, ε, έχουμε βελτιώσει ε, οι εμπορικέ συμφωνίε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κατάσταση των Ιρανών. Υπάρχουν, θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε έως, έως ότου ε, πετύχουμε θετικά και συγκεκριμένα αποτελέσματα όσον αφορά για παράδειγμα την βελτίωση της θέσης των ε, γυναικών. Ο κύριος Ούρμπαν Κρέσπο, ευχαριστώ κυρία Μογκερίνη. Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο εκτέλεσε τουλάχιστον 2.200 ανθρώπους την τελευταία δεκαετία και δεν είχαν επαρκή νομική βοήθεια, υποχρεώθηκαν να υπογράψουν έγγραφα και ομολογήσεις που δεν καταλάβαιναν. Ο αριθμός των κατηγορουμένων έχει εκτοξευθεί σε αστρονομικά επίπεδα από τότε που ο βασιλιάς Σαλμάν ανέβηκε στο θρόνο πέρσι τον Ιανουάριο. Και τώρα φαίνεται να έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα εσείς είχατε τη Σαουδική Αραβία ως προτιμόμενο εταίρο και συνεργάτη στην περιοχή χάρη στις πλούσιες συμβάσεις ε, για τις γερμανικές, γαλλικές, βρετανικές και ισπανικές εταιρείες εξαγοράστηκαν ε, και σιώπησαν ενώ παρίσταντο στην καταστρατήγηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν εξαγορεστεί συνειδήσεις κυβερνήσεων και άλλων και όλα αυτά τα μάθαμε από το Wikileaks. Η Σαουδική Αραβία μπήκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών χάρη στη στήριξη της Βρετανίας, αν είναι δυνατόν. Κυρία Μογκερίνη, με αυτούς τους εταίρους των ευρωπαϊκών πολυεθνικών το μόνο που θα κάνει είναι να αναζωπυρώνεται η φωτιά και δεν θα δοθεί ένα τέλος στους θανάτους. Αποφασίστε. Θα συνεχίζετε να δίνετε βραβεία Ζαχάροφ στους ακτιβιστές της Σαουδικής Αραβίας και από την άλλη να κάνετε το πάνε έτσι ώστε οι εταιρείε να παίρνουν συμβόλαια. Ε, στη Σαουδική Αραβία και στο Ιράν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σμίθ παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Μογκερίνη, είστε ευπρόσδεκτοι πάντοτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλωσορίζω την πρόοδο που έχει γίνει στο Ιράν και προσδοκώ να καλωσορίσω τη χώρα αυτή που θα επιστρέψει από το κρύο. Μπορούμε να συνεργαστούμε με τις δημοκρατικές δυνάμεις και συνεχίστε παρακαλώ τις προσπάθειές σας. Ωστόσο, ενώ προοδεύουμε με την Τεχεράνη, στη Σαουδική Αραβία υπονομεύεται η κατάσταση. Υπάρχει καταστολή στο εσωτερικό της χώρας, υπάρχει αύξηση της κρίσης, καταστροφικές στρατιωτικές παρεμβάσεις στο εξωτερικό, π.χ. η Εμένη. Δύσκολη είναι η προσέγγιση αυτή. Σε κάθε περίπτωση το Ηνωμένο Βασίλειο από το 2010 έχει πουλήσει όπλα αξίας 5,6 ε, ε, δισεκατομμυρίων. Έχουμε την οργάνωση «Σώστε τα παιδιά στην Ιεμένη». Δίνεται η εντύπωση ότι οι πωλήσει όπλων ουσιαστικά διακινδυνεύουν τις ζωές των παιδιών. Βλέπετε πόσο η κριτική μας έχει ασκηθεί. Πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα, κυρία Μοκερίνη, και θα σας το απευθύνω και γραπτός αύριο. Είναι αρκετά αμφισβητούμενη η νομιμότητα των διεθνών συμφωνιών πωλήσεων όπλων. Ειδικά όταν χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στην Ιεμένη. Έχετε αξιολογήσει ε, την νομιμότητα και αν όχι, μήπως δεν θα πρέπει να το κάνετε. Μήπως θα πρέπει να το κάνετε. Ευχαριστώ. Κύριος Καστάλντο, Ξέρετε ότι ορισμένοι συνομιλητές θεωρούνται πιο ισότιμοι από κάποιους άλλους, ιδίω αυτοί οι οποίοι έχουν πετρέλαιο και μπορούν να επενδύσουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια μέσω του πετρελαίου και το είχε πει αυτό και ο Τζορτζ Όρουελ όταν αναφερόταν στις πολιτικές ελευθερίες στον κόσμο και αναφερόμενο στις εξτρεμιστικές δυνάμεις καθώς επίσης και στον πόλεμο τον οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή να εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Κλιμάκωση της βίας χωρίς προηγούμενο. Εμείς πώς αντιδρούμε αυτή τη στιγμή. Θα τρομάξουμε τη Σαουδική Αραβία προκειμένου να αλλάξει στάση. Θα ασκήσουμε πίεση μέσω του πετρελαίου, μέσω της μείωσης της τιμής του ή της μείωσης της παραγωγής. Ή θα ζητήσουμε από τους συμμάχους μας να συνταχθούν όλοι με τις Ηνωμένε Πολιτείες προκειμένου τελικά να ακολουθήσουμε και σε Σαουδική Αραβία μια συμφωνία στην αυτή που είχαμε με την πυρηνική ενέργεια στο Ιράν Νομίζω ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει να δούμε ότι όλοι οι σύμμαχοι θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι κατά της τρομοκρατίας, κατά όσων χρηματοδοτούν την τρομοκρατία ή υποστηρίζουν την τρομοκρατία, αλλά κατά και αυτών που προωθούν τη θανατική ποινή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουν ορισμένα κράτη-μέλη ότι έχουν και αυτά προωθήσει πάρα πολλά όπλα προς τις χώρες, τις περιοχές, στην περιοχή αυτή. Και καταλαβαίνετε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να πειράσουμε περισσότερο περισσότερο θετικά τα πράγματα και να αποφύγουμε την κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ιεμένη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η σύγκρουση μεταξύ Σαδικής Αραβίας και Ιράν ε, ε, ενέχει τον κίνδυνο να μπει σε μια καυτή ε, φάση. Και ε, μια τέτοια σύρεξη θα οδήγησει ολόκληρη την περιοχή σε όλεθρο και αυτό θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις και για την, Ευρωπαϊκή, για την Ευρώπη. Και χαιρετίζω το γεγονός ότι το Εράν μετά την ε, ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την πυρηνική ε, περνάει σε μια νέα φάση. Ε, κανείς ε, δεν μπορεί να ενδιαφέρεται σε μια αποσταθεροποίηση στην ε, περιοχή. Όλες οι δραστηριότητες που έχουν σαν στόχο με την υποστήριξη του Ισλαμικού κράτους να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή είναι επικίνδυνες. Η σταθερότητα δεν επιτυγχάνεται με την καταστολή αλλά μακροπρόθεσμα επιτυγχάνεται μέσω του κράτους δικαίου. Ε, η Σαουδική Αραβία δυστυχώς ε, απέχει παρασάγκασα από αυτές τις εξελίξεις και αυτό το κατέδειξαν και τα τελευταία γεγονότα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε προς τα που κατευθύνεται η Σαουδική Αραβία. Ε, θα πρέπει ωστόσο εμείς από την πλευρά μας να περιορίσουμε τις δικές μας προμήθειες όπλων προς την Σαουδική Αραβία. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε το λόγο. Ο στόχο τη πολιτική μα θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση τη ειρήνη και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Εγγύη Ανατολή. Η εξέλιξη στην περιοχή αυτή, ειδικά για μα στην Ευρώπη, είναι μεγάλη σημασία γιατί ε, από τη Συρία αλλά και από αυτές τις περιοχές προέρχονται οι περισσότεροι πρόσφυγες. Ωστόσο γεγονό είναι ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο στη Σαουδική Αραβία όσο και στο Ιράν ε, παραβιάζονται κατάφορα, ποδοπατούνται θα έλεγα και οι δύο χώρες εμπλέκονται σε πολέμους όχι μόνο στην Ιεμένη αλλά η Σαουδική Αραβία έμεσα μέσω χρηματοδότησης στη Συρία και το Ιράκ αυτή τη στιγμή όμως εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια δυνατότητα γιατί η Σαουδική Αραβία απομακρύνονται λίγο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πλησιάζουν προς την Ευρώπη και μια αντίστοιχη ευνοϊκή κατάσταση έχουμε και στο Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να επιβάλλουμε ευκολότερα τα δικά μας αιτήματα και ε, βεβαίω ε, αυτό θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βεβαίως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τερματίσει άμεσα την εξαγωγή όπλων στο Ιράν. Κύριος Ποστινάρχη το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπατή Εκπρόσωπε, προφανώς υπάρχει κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο φτωχωρών και αυτό μας ανησυχεί ιδιαιτέρως. Το πρόβλημα αυτό αφορά βέβαια μια περιοχή η οποία ήδη πλήττεται από άλλους πολέμους και άλλες διενέξεις. Ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να συμβάλλει επικοδομητικά και να φέρει στο τραπέζι των πραγματεύσεων και τις δύο αυτές χώρες. Η διαδικασία της Βιέννης για τη Συρία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπονομευτεί και η όλη αυτή περιοχή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει απλώ μια περιοχή αντιπαράθεση και αντιπαλότητα μεταξύ Σουνιτών και Σίτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει επικοδομητικά και να πείσει τις δύο αυτές πλευρές να οδηγηθούν μακριά από οποιαδήποτε κλιμάκωση της βίας. Ο κύριος Τζοφόλ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν άλλαξε εντελώ το τοπίο στη Μέση Ανατολή. Η επιθετικότητα και η εχθρότητα πολλές φορές των Αμερικανών κατά του Ιράν και η φιλία υπέρ της Οδικής Αραβίας αποτελούσε ένα γενικότερο υπόβαθρο των όλων εξελίξεων που είχαμε στη Μέση Ανατολή. Και αυτό που είχαμε δει στο παρελθόν, στην περιφέρεια αυτή, είναι ότι πέρα από το Μεσανατολικό είχαμε μία αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και άλλων χωρών και συγκεκριμένα μεταξύ Σιητών και Σουνιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε λοιπόν να συμβάλλει σημαντικά στην διαπραγμάτευση που έγινε για το πυρηνικό πρόγραμμα για το Ιράν και να ευχαριστήσουμε εδώ πέρα την κυρία Μογκερίνη. Η συμφωνία αυτή που αποτελεί το μόνο ελπιδοφόρο μήνυμα που έχουμε το τελευταίο διάστημα θα πρέπει να οδηγήσει σε καλύτερες διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν και με καλύτερη σχέση της χώρας αυτήν με το Αφγανιστάν, το Ιράκ και θεωρώ ότι θα μπορούσε να υποφελήσει την όλη περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει παράγοντα σταθεροποίηση στην περιοχή και μπορεί να συμβάλλει στο να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία. Δεν θα πρέπει όμω σε καμία περίπτωση να έχουμε εμπριστικέ δηλώσει από διάφορε πλευρέ. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει να θέσουμε εν κινδύνο τη ερευνητική διαδικασία στη Συρία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να, να καταδικάσουμε τη θανατική ποινή. Όσο περισσότερο Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε, τόσο περισσότερο θα ενισχύεται η Ευρώπη, τόσο περισσότερο θα ενισχύεται η Κυρίνη. Η κυρία Γκόμε έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε. Αυτό το οποίο βλέπουμε πάρα πολλές φορές στην περιοχή αυτή είναι ότι υπάρχουν διάφοροι ηθήνοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην κλιμάκωση της βίας. Πρέπει να ακολουθήσουμε, όπως είπαν και οι προαλήσαντες, την ε, διαδικασία της Βιέννη οι Ιρανικές ε, αρχές Ξέρετε ότι πολλές φορές έχουν ακολουθήσει ακραία στάση. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε πλέον μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Έχουν αρθεί οι κυρώσεις. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να συμβάλλουμε σε μια ειρηνευτική διαδικασία, κυρία Μογκερίνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικρίνει όποτε κρίνεται αναγκαίο το Ιράν, ιδίω για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα όμω θα πρέπει να συνεργαστούμε και με το Ιράν ένα κράτος το οποίο λειτουργεί στην πράξη και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε τέλος στον πόλεμο της Συρίας και θα καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε κάθε τρομοκρατική οργάνωση συμπεριλαμβανομένου του Ισλαμικού κράτους. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να συμβάλλουμε θετικά στην όλη περιοχή. Η κυρία Μόσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την ύπατη εκπρόσωπο γιατί αναφέρθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση που υπάρχει μεταξύ Σαουδική Αραβία και Ιράν. Μας ανησυχεί και εμά ιδιαίτερα η κατάσταση αυτή, ιδίω από το φω τη συζήτηση που μόλι τώρα ολοκληρώσαμε, ιδίω όσον αφορά την ερευνητική διαδικασία για την Συρία και ιδίως υπό το φω των τελευταίων εξελίξεων που είχαμε, όπου είδαμε τελικά ότι στο διάλογο τον ειρηνευτικό πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αποκλείσουμε λοιπόν τη συνεργασία και με τις δύο αυτές πλευρές, και με τη Σαουδική Αραβία και με το Ιράν. Επίσης σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θέσουμε εν κινδύνο το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα το οποίο είχαμε στο Ιράν με το πυρηνικό πρόγραμμα. Τέλος, Χαιρόμαστε πάρα πολύ που αναφερθήκατε, κυρία Μογκερίνη, στι συνεχεί προσπάθειε που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάργηση τη αντική ποινή και για το γενικότερο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Δεν είναι πουσιώδη τα ζητήματα αυτά. Θα πρέπει να αποτελέσουν απόσπαστο τμήμα οποιασδήποτε στάσει έχουμε απέναντι σε οποιονδήποτε διεθνή εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μαμίκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Μογκερίνη, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι τελευταίες εξελίξεις αποσταθεροποιούν την Μέση Ανατολή. Η εκτέλεση του Σεΐχη, του Σιήτη Σεΐχη ήταν ανεύθυνη πράξη από τη Σαουδική Αραβία. Το Ιράν θέλησε να προστατεύσει την πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας και γι' αυτό διάκοψε τις διπλωματικές σχέσεις. Ωστόσο αυτή είναι μια δυσανάλογη απάντηση. Υπάρχει διαφορετικός δρόμος να εφαρμοστεί η συμφωνία με το Ιράν, να αρθούν οι κυρώσεις και έτσι θα συνεργαστούμε επικοδομητικά. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε από τη Συρία. Οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας δεν πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο τις ειρηνευτικές συνομιλίες στη Συρία. Όπως έχουν αποφασιστεί από το ψήφισμα του ΟΗΕ, καλό αμφότερες πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα. Και θέλω να τονίσω ότι για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης θα πρέπει η Σαουδική Αραβία να σταματήσει τη χρηματοδότηση των εξτρεμιστών που διέπονται από γουαχαβητική ιδεολογία και που ευθύνονται για τους διαφόρους βομβαρδισμούς και επιθέσεις στην Αίγυπτο, στο Παρίσι και αλλού. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, ε στη διαδικασία Catch the Eye, γιατί είναι αργά. Ο κύριος Πόλτσακ καταρχάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου στα βήματα της κυρίας Μογκερίνη. Τα βήματα που κάνει είναι συνεκτικά, συνεπή, τα έχει σκεφτεί σωστά. Ποια απόφαση λάβατε το Σάββατο τι περιλαμβάνει, τι σημαίνει για παράδειγμα για την αντιπολίτευση στη Σαουδική Αραβία. Τι σημαίνει για όλους αυτούς που εκπροσωπούν την αντιπολίτευση στη Αραβία, οι οποίοι νιώθουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ξέχασε. Πιστεύω και ελπίζω να μην είναι έτσι. Θα στηρίξουμε τα μέρη της κοινωνίας, τα τμήματα της κοινωνίας που προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό και η αποκλιμάκωση που ανέφερε η κυρία Μογκερίνη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ελπίζω η συνεισφορά μας να διαρκέσει σε αυτή την περιοχή την τόσο ευπαθή. Ευχαριστώ. πρόεδρε, τα πρόσφατα συμβάντα στη Σαουδική Αραβία και στο Ιράν ε, ε, αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ανησυχώ εάν, για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν πάρει θέση ε, σε αυτή τη σύγκρουση θα επιδεινώσει τις εξελίξεις και αυτό θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις ε, στην Συρία αλλά και στην Ιεαμένη και ενδεχομένω θα πυροδοτήσει συγκρούσεις σε άλλα μέρη του κόσμου. Ωστόσο υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι μπορεί να γίνει το για την Μέση Ανατολή. Θα ε, χαιρετίζω την άρση των κυρώσεων και θα χαιρέτησα επίσης μια χρηματοδότηση η οποία θα βελτιώσει τις συνθήκε διαβίωσης των ε, πολιτών. Ε, μου έκανε εντύπωση για η εκλογή της πρώτης ε, γυναίκας ε, πολιτικού στη Σαουδική Αραβία. Και δύο πλευρές θα πρέπει να τηρούν την αρχή της μη παρέμβασης σε κυρίαρχα κράτη. Uh, Ευχαριστώ. Εντός του Ισλάμ υπάρχει μια διαφορά μεταξύ Σουνιτών και Σιητών. Υπάρχουν περαιτέρω διαφορές εντό ε, των ε, Σουνιτών αλλά η εξαγωγή της ε, ιδεολογίας, ε, της ιδεολογίας αυτής οδηγεί στην ενίσχυση των δογμάτων του ίσης ε, το ίσης φωνεύει όλους όσοι είναι χριστιανοί, νομοφιλόφιλοι κλπ. Ε, Ωστόσο, Βρετανοί συνάδελφοι δεν υπερασπίστηκαν αυτή τις θέσεις. Πολλοί πιστεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Μογκερίνη, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Να πω καταρχάς ότι α, ε, όντως υφίσταται, όπως υπήρχε πάντα, ένας διαχωρισμός μεταξύ Σουνιτών και Σιητών, αλλά διαχωρισμοί υπάρχουν και μεταξύ των ίδιων των Σουνιτών. Και σίγουρα τα πράγματα είναι αρκετά πολύπλοκα και στην περιοχή και πέρα από την περιοχή. Και κάτι ακόμα. Κάτι το, με το οποίο συμφωνούν πάρα πολλοί φίλοι και τέρημα στην περιοχή. Ότι η διαχωρισμοί και την παράθεση δεν είναι τόσο θρησκευτική φύση, αλλά πολιτική κυρίω φύση. Μια πολιτική αντιπαράθεση που χρησιμοποιεί ω πρόσχημα τη θρησκεία τελικά. Και οι Σουνίτες και οι Σίτες βέβαια σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, αλλά ακόμα και στο Ιράν, ζούνε στο Ιράκ με συγχωρείτε, ζουν ειρηνικά μαζί. Και αυτό έγινε ή γινότανε πρωτοί πολιτικοποιηθεί αυτός ο σεχταριστικός διαχωρισμός που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ο δικός μας λοιπόν ο ρόλος θα μπορούσε να ήταν να διευκολύνουμε ευρύτερες επενδύσεις σε αυτό το οποίο ορισμένοι είπατε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια συλλογική αρτεκτονική ασφάλεια στην όλη περιοχή. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εγγυηθούμε την ειρήνη και την ασφάλεια σε μια περιοχή που είναι πάρα πολύ σημαντική για τον υπόλοιπο κόσμο. Και ακριβώ επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα επαρκέ όραμα μια συλλογική αρχιτεκτονική ασφάλεια, βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε και έχουμε την κλιμάκωση τη βία που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα εμεί για να βοηθήσουμε την κατάσταση. Κάτι το οποίο είναι προ το συμφέρον μα προφανώ. Πρώτον, και το είπατε ορισμένοι από εσά, α μην ταχθούμε με τη μία ή την άλλη πλευρά έχουμε καλές ή σχετικά καλές τουλάχιστον σχέσεις, σχέσεις εργασίας, ανοιχτές διάβλους, οι οποίες λειτουργούν τις περισσότερες φορές και με το Ιράν και με την Σαουδική Αραβία. Και προφανώς η εφαρμογή της συμφωνίας που υπογράψαμε το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα μπορεί να οδηγήσει και σε νέες ευκαιρίες για τις διμερείς σχέσεις που έχουμε με το Ιράν. Έχουμε λοιπόν σχέσεις και με το Ιράν και με τη Σαουδική Αραβία, τις οποίες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έχοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να είναι σαφείς προς όλους τους εταίρους και τους εμπλεκόμενους στην περιοχή. Μία ατζέντα προτεραιότητες οι οποίες περιλαμβάνουν προφανώς την αντιμετώπιση της διμερούς αυτής αντιπαράθεσης, τη χρησιμοποίηση της περιφερειακής δυναμικής που υπάρχει, το γεγονός ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε πολιτικές λύσεις για όλες τις διενέξεις που έχουμε στην περιοχή, ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την αθεκτικότητα κάποιων βασικών κρατών, οι οποίες, ε, τα οποία κράτη με συγχωρείτε εκτίθενται στην ε, βία αυτή, Ιράκ, Λίβανος κτλ και βέβαια θα πρέπει να δούμε και ποιε είναι ιστορικέ εξελίξει χώρε αυτέ και ποια είναι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητήματα τα οποία πάντα συζητούμε και με τη Σαουδική Αραβία και με το Ιράν. Και να απαντήσω σε όσους ε, αναφέρθηκαν στο ζήτημα του πετρελαίου. Ενδεχομένω θα πρέπει λίγο να ξαναδείτε τα πράγματα γιατί ε, η τιμή του πετρελαίου που έχουμε αυτή τη στιγμή παγκοσμίω τροποποιεί εντελώ τι σχέσει που έχουμε με τι χώρε αυτέ και με τι χώρε του κόλπου. Επομένω, έχουμε μια ξεκάθαρη πολιτική ατζέντα, ξεκάθαρε πολιτικέ προτεραιότητε και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια προνομιακή θέση αυτή τη στιγμή κάθε φορά που συνομιλούμε με τέρους στην περιοχή. Γιατί όπως σας είπα δικές μας οι προτεραιότητες είναι συνεκτικές και σαφείς. Και ναι, όντω. Υπάρχουν πολλές φορές αποκλίνουσες προτεραιότητες μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγχωρείτε, αποκλίνουσε ατζέντε οικονομικέ μεταξύ διαφόρων κρατών τη περιοχή, αλλά εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση κινούμαστε ενωμένοι. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να επενδύουμε περισσότερο στην καλλιέργεια των σχέσεων αυτών με το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία, με τον λαό των κρατών αυτών, με κάθε δυνατή μορφή και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για δύο βασικούς στόχους εξωτερικής μας πολιτικής. Από τη μία πλευρά τον έχουμε ένα πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και δεύτερον κάτι το οποίο αποτελεί ε, σημαντική προτεραιότητα και με τη Σαουδική Αραβία και με το Ιράν και με άλλες χώρες το ότι ε, δίνουμε μάχη για την καταπολέμηση και την ε, κατάργηση της θανατικής ποινή παντού στον κόσμο, βασιζόμενη στις αρχές μας, στα πιστεύω μας, αλλά και στην εμπειρία μας, διότι γνωρίζουμε ότι η θανατική ποινή δεν είναι αποτελεσματική. Προφανώς είναι απάνθρωποι, αλλά δεν είναι καν αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν για την ε, η υποστήριξή σας προς ε, τη δράση που έχουμε αναλάβει στο ζήτημα αυτό. Η υποστήριξή σας θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και στο μέλλον και για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ για όλη τη συμβολή σας, την εργασία που έχουμε καταβάλει εμείς για την όλη αυτή περιοχή που είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά την ασφάλεια και τη σταθερότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μογκερίνη.